σχετικά με τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης της 17 η ε, Ιανουαρίου τα έχετε στην διάθεσή σας και περνάμε τώρα στις ε, ανακοινώσεις του Πρόεδρου.